Και τώρα περνάμε στην ημερήσια διάταξη. Το οριστικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης που εγκρίθηκε από τη διάσκεψη των Προέδρων στις 11 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το άρθρο 149, σας έχει διανεμηθεί. Η ημερήσια διάταξη λοιπόν θεωρείται ότι εγκρίνεται. Και περνάμε στην Δευτέρα, δηλαδή σήμερα. Η Γκουε έχει ζητήσει να αναβληθεί η συζήτηση και η ψηφοφορία για την έκθεση του κυρίου Μάτο μετά από αυτή την απόφαση παρακαλώ με τον τίτλο «Διατήρηση των αλλιευτικών πόρων και προστασία των ε, θαλασσίων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων». Αυτό το αίτημα στηρίζεται από την ομάδα των Πρασίνων και από την EFTD. Δίνω το λόγο στον κύριο Μαρή για να ε, διατυπώσει την, ε, το αίτημα της ΓΚΟΕ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, η ομάδα μας ζητά όντως την αναβολή της ψηφοφορίας για την έκθεση του συναδέλφου Καμπριέλ Μάτο για πολλούς λόγους ε, ε, αλλά θα σας αναφέρω μόνο έναν, ότι δηλαδή πριν λίγες μέρες ο τύπος και η ΜΚΙΟ αποκάλυψαν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε λάβει υπόψη τα συμπεράσματα μιας έκθεσης εμπειρογνωμόνων που ωστόσο η ίδια είχε ζητήσει αυτή την έκθεση, μια έκθεση που, που κατέληγε ε, στο πόσο επικίνδυνη είναι ε, το ηλεκτρικό, το, το, το ψάρεμα μέσω του ηλεκτρισμού. Ωστόσο, η Κομισιόν στην έκθεση αυτή λέει το αντίθετο από αυτό που έλεγε η έκθεση των εμπειρογνωμόνων και ε, που έλεγε δηλαδή ως κατάληξη ότι πρέπει να απαγορευτεί αυτού του είδου η βάρβαρη αλληλεία. Η Κομισιόν λοιπόν έχει θελημένα ε, πει ψέματα στους ευρωβουλευτέ. Αυτό είναι το ερώτημα και αυτό είναι το ερώτημα που οφείλουμε να τη θέσουμε πριν να μπορέσουμε να λάβουμε θέση νυφάλια και γνωρίζοντα πλήρως το θέμα για μια ανέκθεση που αναμένεται όλος ιδιαίτερος και επί της οποίας το Ευρωκοινοβούλιο καλύτερα να αποφασίσει. Και γι' αυτό και σας ζητώ να υπερψηφίσετε την αναβολή της ψηφοφορίας για αυτήν την έκθεση. Κύριε Φερχόφστατ, θέλετε να μιλήσετε ενάντια σε αυτή την πρόταση. Όχι, για διαδικαστικό θέλω να το λόγο το θέμα αυτό, επειδή υπήρχαν πάνω από 200 τροπολογίες και χωριστές σοφορίες και το άρθρο 175 του κανονισμού δίνει την δυνατότητα, αν υπάρχουν τόσες τροπολογίες και τόσο μεγάλη αβεβαιότητα, να αναπαιμφθεί στην Επιτροπή. Και η πρότασή μου είναι να εφαρμόσετε το άρθρο αυτό, το 175 του κανονισμού, λόγω του πληθωρισμού ε, τροπολογιών και να την αναπέμψετε στην Επιτροπή. Και έτσι θα υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει κάποια σαφήνεια και αντικειμενικότητα στο θέμα αυτό, γιατί έχω, την... έχω μια περίεργη αίσθηση εδώ πέρα ότι διαβάζουμε επιστημονικά στοιχεία υπέρ της μίας και της ακριβώς αντίθετης θέσης. Και δεν είναι φυσιολογικό. Κανονικά υποτίθεται ότι στην επιστήμη υπάρχει μία αντικειμενικότητα. Προτείνω λοιπόν να το ε, ξαναστείλετε στην Επιτροπή με βάση το άρθρο 175 για να ξεκαθαρίσει το ζήτημα για να υπάρξει μία πιο αντικειμενική εξέταση ε, από το να το ψηφίσουμε αύριο εδώ στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Φερχόφστατ που μου θυμίσατε αυτή την δυνατότητα. Κύριε Μάτο, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, όντως, πρέπει να βλέπουμε τι είναι λογικό και τι είναι παράλογο. Εδώ λοιπόν έχουν τεθεί δύο διαφορετικά ζητήματα. Το πρώτο είναι το θέμα του εισαλληλίας ε, με τον ηλεκτρισμό. Ε, θα πρέπει να σας θυμίσω ότι εργαζόμαστε για αυτό το θέμα εδώ και 21, 21 μήνες. 77 ε, αναφορές έχουν γίνει αιτήματα για να τεθεί αυτό το θέμα στην Ολομέλεια τον Ιούνιο. Την αναβάλαμε για τον Σεπτέμβριο, την αναβάλαμε και για τον Οκτώβριο. Προτάθηκε να συζητηθεί, να ψηφιστεί το Δεκέμβριο. Κάποιος πρότεινε να αναβληθεί για σήμερα και, την αναβάλαμε λοιπόν για σήμερα. Ποτέ κανεί δεν ανέθεσε αυτό το πρώτο θέμα, αυτό που τίθεται σήμερα, δηλαδή το θέμα τη ε, αλληλεία με, με ηλεκτρισμό. Και, όμως αυτό το οποίο τίθεται αυτή τη στιγμή είναι ότι δηλαδή ε, το 2006 η Κομισιόν, δηλαδή πριν 12 χρόνια, ε, ήρε μια απαγόρευση. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να το συζητήσουμε σήμερα και να το ψηφίσουμε αύριο. Εάν, όπως είπε ο κύριος Μάρζε, ότι αυτό το θέμα είναι, για, είναι προς απαγόρευση, ε, θα πρέπει να το δούμε. Ε, δεν πρέπει τώρα να χρησιμοποιήσουμε αυτήν εδώ την ευκαιρία για να ε, τιμωρήσουμε την Κομισιόν επειδή έκανε κάτι το 2006. Επιπλέον, εάν επανέλθει το θέμα αυτό στην Επιτροπή, 92, 92 ε, τροπολογίες Ορισμένες από αυτές έλαβαν πάνω από το 1 τρίτο των ψήφων, ε, θα διατηρηθούν και για την Ολομέλεια. Αυτό σημαίνει ότι 80% περίπου των τροπολογιών έχουν εγκριθεί ή έχουν απορριφθεί ίσα ίσα, με σχεδόν ισοψηφία. Σε κάθε περίπτωση αυτές οι τροπολογίες θα ξαναέρθουν στην Ολομέλεια γιατί θα ξεπεράσουν το 1 τρίτο των ψήφων. Δηλαδή δεν θα καταφέρουμε τίποτα ακόμα και αν το αναβάλουμε. Αυτή η δικαιολογία χρησιμοποιήθηκε ώστε ορισμένε ομάδες που δεν συμφωνούν με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στην αρμόδια επιτροπή χρησιμοποιείται για να προσπαθήσουν να αλλάξουν κάπως τις ισορροπίες. Δεν υπάρχει όμως τίποτα το νέο για τα όσα έχουν προταθεί και δεν υπάρχει λόγος να αναβληθεί πάλι το κείμενο. Εγώ προτείνω να διατηρηθεί η συζήτηση και να ψηφίσουμε αύριο. Θα αποφασίσει λοιπόν η Ολομέλεια που έχει και την ε, αρμοδιότητα. Ψηφίζουμε για την πρόταση της ομάδας Γκουε να αναβληθεί η ψήφιση της έκθεσης ε, ΜΑΤΟ για την, ε, για την ηλεκτρικών μέσων και τη χρήση τεχνικών μέτρων και την προστασία των θελάσσιων πόρων. Άρχεται η ψηφοφορία.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 Απορρίπτεται η πρόταση. Οπότε και συζήτηση θα γίνει και θα ψηφιστεί εφόσον η πλειοψηφία αποφάσισε έτσι. Σε ό,τι αφορά την τρίτη, η ομάδα Γκουε ζήτησε ως τέταρτο σημείο στην ημερήσια διάταξη να περιληφθεί το απόγευμα ένα προφορικό ερώτημα σε σχέση με την συνθήκη για την απαγόρευση το χρήσης πυρηνικών όπλων. Ο λόγος στον κύριο Βιέγκας για να αναπτύξει την πρόταση της ομάδας του. Το θέμα των πυρηνικών όπλων είναι ε, ιδιαίτερα επίκαιρο. Στην ημερήσια διάταξη έχουμε όλο και μεγαλύτερη ένταση και στον ΟΗΕ συζητείται ένα δεσμευτικό μέσο, ένα δεσμευτικό εργαλείο υπό τη μορφή μια συνθήκη για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ολομέλη να συζητήσει αυτό το ζήτημα. Πρόκειται για την παγκόσμια ειρήνη και εν τέλει η ίδια η επιβίωση του πλανήτη μας. Προτείνουμε λοιπόν η συζήτηση να γίνει την Τρίτη το απόγευμα γύρω από την προφορική ερώτηση που θέσαμε στο Συμβούλιο και ζητάμε επίσης η ψηφοφορία για αυτή την πρόταση να γίνει με ονομαστική κλίση. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Θέλει κανείς να εκφράσει αντίθετη άποψη. Παρακαλώ, κύριος Λάμπερτς. Κύριε Πρόεδρε, Πιστεύω ότι το, θέμα των πυρηνικών όπλων φυσικά και είναι χρήσιμο. Θέλω απλά να πω ότι βεβαίω εάν υποστηρίζουμε την ιδέα να το συζητήσουμε εδώ, νομίζω πω δεν έχουμε κάτι νέο από τη διάσκεψη του Πρόεδρου τη περασμένη Πέμπτη, όπου να πρέπει δηλαδή επιγόντως να το συζητήσουμε. Πιστεύω πως θα ήταν πιο φρόνιμο να το συζητήσουμε το Φεβρουάριο, δηλαδή να προετοιμαστούμε καλύτερα και να το συζητήσουμε το Φεβρουάριο. Είμαστε υπέρ του να συζητήσουμε αυτό το θέμα στην Ολομέλεια. Μάλιστα. Αν κατάλαβα καλά κύριε Λάμπρες, εσείς προτείνετε να συζητηθεί αυτή, αυτό το θέμα το Φεβρουάριο και όχι τώρα. Εσείς επιμένετε στην πρότασή σας. Ναι. Η πρόταση αυτή δεν είναι νέα, ε, την έχουμε ήδη κάνει και γι' αυτό και επιμένουμε στο να συζητηθεί αύριο το απόγευμα το θέμα. Ωραία λοιπόν, ψηφίζουμε με ονομαστική κλίση μετά από αίτημα της ομάδας ΓΟΕ να προσθέσουμε ως τέταρτο σημείο στην σε διάταξη αύριο το απόγευμα μια προφορική ερώτηση για την συνθήκη για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η πρόταση. Οπότε η μερίσια διάταξη παραμένει απαράλλακτη. Δε Μεσμέκερ έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε επί της ε, διαδικασίας με βάση το άρθρο 151 του κανονισμού. Κύριε Πρόεδρε, στις 19 Δεκεμβρίου κάποιοι συνάδελφοι μεταξύ των οποίων και εγώ θέλαμε να επισκεφθούμε την φυλακή Εστρεμέρα ε, κοντά στη Μαδρίτη όπου κρατείται ο πρώην συνάδελφός μας Ριόν Σουνκέρας. Ε, ε, πρόκειται λοιπόν για δύο ηγέτες και δύο πρώην υπουργούς του καταναλανικού κινήματος και βεβαίως είχα μαζί μας ε, και βουλευτές ε, του Κοινοβουλίου της ε, Καταλωνίας και ζητούσαμε επί ένα μήνα να μας επιτραπεί η επίσκεψη. Τώρα λάβαμε μια επίσημη απάντηση. Όταν φτάσαμε εκεί μας αρνήθηκαν την είσοδο και δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε και με τον διευθυντή καν της φυλακής. Πρόκειται για απαράδεκτο τρόπο λειτουργίας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συχνά διαμαρτυρόμαστε όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο στην Τουρκία ή σε άλλες τρίτες χώρες. Θεωρείτε κύριε Πρόεδρε ότι οι Ισπανικές αρχές ε, θα πρέπει τουλάχιστον να δώσουν εξηγήσει ή θα πρέπει να διαμαρτυρηθούμε επισήμως. E θα κοιτάξουμε κατά πόσο υπόθηκε αυτό και την Πέμπτη, κατά τα άλλα, η ομάδα ΓΚΟ έχει προτείνει να προσθεθεί ω δεύτερο σημείο στην μεσαδιαταξή η δήλωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι μαζικέ απολύσει σε ανταγωνιστικέ επιχειρήσει στην Ευρώπη και την υπόθεση Siemens. Ο λόγο στον κύριο Σέρντεβαν για να διατυπώσει την πρόταση τη ομάδα του. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η Siemens ΑΕ παρά τα τεράστια κέρδη της ανακοίνωσε κλείσιμο εργοστασίων και απολύσεις. 7.000 απολύσεις ε, κυρίως αφορούν Ολλανδία και Γερμανία χωρίς να μετράμε τους ανθρώπους ε, σε επιχειρήσεις που προμηθεύουν την ε, Siemens ε, και μιλάμε για την μοίρα ολόκληρων ευρωπαϊκών περιφερειών που απειλούνται από τις περιοχές παρά το ότι τα εργοστάσια αυτά είναι κερδοφόρα παρά το ότι η Siemens στην ε, Γερμανία είχε λάβει 300 εκατομμύρια ευρώ κρατικές ενισχύσεις. Αυτό για την ομάδα μας, ε, την QNGL, αρκεί για να ζητήσουμε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Ζητώ τη συμφωνή σας γνώμη για να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης ε, στους εργαζόμενους αυτούς και να πούμε ότι δεν επιτρέπεται να κάνουν μαζικές απολύσεις κερδοφόρες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Ποιος θα τοποθετηθεί κατά της συμπεριλήψη στην ημέρα διάταξη αυτού του σημείου προ συζήτηση. Εάν κανεί δεν θέλει να πάρει το λόγο, να ψηφίσουμε με ονομαστική ψηφοφορία για την πρόταση τη ομάδα ΓΟΕ να προσθεθεί ω δεύτερο σημείο στην ημερήσια διατάξη τη 5η το πρωί η δήλωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τι μαζικέ απολύσει σε ανταγωνιστικέ επιχειρήσει στην Ευρώπη και την περίπτωση Siemens. Η ψηφοφορία άρχεται τώρα. avete votato tutti onorevole mcallister bene allora la Ωραία. Η ψηφοφορία έληξε. Η πρόταση απορρίφθηκε. Η ημερήσια διάταξη παραμένει ως έχει. Έχει λοιπόν αποφασιστεί και εγκριθεί. Περνάμε στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, κοινή συζήτηση για την καθαρή ενέργεια με τις εκθέσεις Μπλάνκο Λόπες, Ποχ, Ριβαζή και Τούρμες. Πρώτος ο κύριος Μπλάνκο Λόπες, ως αρμόδιος εισηγητής.